Προσοχή, ξεκινάμε 8.30 αύριο, 18 Απριλίου και η μερίσια διάταξη δημοσιεύθηκε και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Διακόπτουμε για την ώρα και καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.